Ας αρχίσουμε με τις ε, επεξηγήσεις ψήφου, παρακαλώ. Έχουμε πρώτα απ' όλα την έκθεση Γκραφ ε, ο κύριος Χάνανα. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Ελβετία, η Ελβετία, μια εύπορη, επιτυχημένη φιλενική χώρα, υψηλό επίπεδο δημοκρατικής ικανοποίησης, υψηλότατα πρότυπα βάση το ΙΕ και φιλικές σχέσεις ε, με τις γειτονικές χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία είναι εταίρος και φίλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διημερίες επίπεδο έχει αναλάβει δεσμεύσει αλλά και διατηρεί για τη διακριτική ευχέρεια να νομοθετεί. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό για όλους όσους δεν είναι δεν υπάρχονται στην αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά μπορούμε να λειτουργούμε ω κυρίαρχα κράτη, όχι ότι θα του αντιγράψουμε. Μπορούμε για τον ΝΑΤΟ, παραδείγματο, να συμμετέχουμε στην ε, άμυνα τη Ευρώπη. Έχουμε ένα κομμάτι τη ενιαία αγορά, αλλά είμαστε εκτό τη πολιτική ένωση. Επιδιώκουν ε, με μεγαλύτερη ολοκλήρωση, διατηρώντα όμω την κυριαρχία του. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο μοντέλο και για άλλε ευρωπαϊκέ χώρε μπορούσε. Ευχαριστώ, Μπαστιά. Σεμπαστιά. Ψήφισα κατά αυτής της ε, καινούργια οικονομικής συμφωνίας ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής και των χωρών ΣΟΕΣ ε, γιατί πλήττει ε, τους παραγωγούς εσπεριδοειδών και, παραγω... και πορτοκαλιών ε, ιδιαίτερα στη Βαλένθια. Η... Τα πορτοκάλια της από την Νότια Αφρική θα μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλήγμα στους παραγωγούς μα γιατί θα συμπίπτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα δικά μας πορτοκάλια με τα εισαγόμενα. Είναι ένα ακόμα χτύπημα στους παραγωγούς πορτοκαλιών ε, που πλήττονται από ε, τον ε, ανταγωνισμό, αθέμητο ανταγωνισμό από τους παραγωγούς της Βόρειας και τώρα και της Νότιας Αφρικής. Ένα ακόμα πλήγμα το οποίο θα ενισχύσει τον ευρωσκεπτικισμό. Πώς θα το εξηγήσω εγώ αυτό στους ψηφοφόρους μου. Μας δίνει την εντύπωση η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν εργάζεται για τα συμφέροντα των δικών μας παραγωγών. Ε, Κυρία Γέρα Γκαρσία. Ψήφισα όχι καταψήφισα δηλαδή αυτή τη συμφωνία γιατί μία ακόμα φορά η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιβαίνει με την κοινή αγροτική πολιτική και ιδιαίτερα αντιβαίνει με τα συμφέροντα των παραγωγών και ιδιαίτερα των σπεριδοειδών. Εγώ προέρχομαι από το νότιο της Ισπανίας, από την Ανταλουσία, ε, όπου όπως και στην ε, Βαλένθια παράγουμε πολλά σπεριδοειδή. Δεν βρήκα καμία ευαισθησία για τα συμφέροντά μας. Επίσης πρέπει να καταγγείλω ότι ο κλάδος αγνούσε πλήρως τις τελευταίες συμφωνίε. τη διεύρυνση κατά έξι εβδομάδες της ε, περίοδου κατά τη διάρκεια τη οποία θα συμπίπτουν οι εισαγωγέ με τη δική μας παραγωγή. Επίση, η πλήρης κατάργηση όλων των δασμών έγινε εναγνία του κλάδου. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να κάνουμε διεθνή εξωτερική πολιτική με τέτοιο τρόπο. Το, η συμφωνία αυτή πλήττει βαριά την ε, κοινοτική μας ε, πολιτική και τους αγρότες μας. Λέω όχι. Κύριε Μακοβέη, την επόμενη δεκαετία οι χώρες της Αφρικής, του Ειρηνικού και της Καραβικής θα απελευθερώσουν το 80% του εμπορίου τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται κατορθωτό μέσω μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης του 2012. Όμως αυτή η συμφωνία δεν είναι πλήρης και δεν είναι και άψογη. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να συνεχίσουμε προκειμένου ε, να συμπεριληφθούν και οι δημόσιες προμήθειες ε, και ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα θέματα και υπηρεσίες. Ε, αυτό θα μας βοηθήσει, αυτή η συμφωνία θα μας βοηθήσει επίσης και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετανάστευσης, διότι η βελτίωση της οικονομίας των χωρών αυτών θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα, το οποίο σημαίνει ότι θα μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Ευχαριστώ. Κύριε Σένρα Ροδρίγες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταψήφισα αυτή τη συμφωνία διότι ε, αντιβαίνει με τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων παραγωγών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε των αγροτών της Νότιας ε, Ευρώπης όσο και των συμφερόντων της Νότιας Αφρικής. Βρισκόμαστε ενώπιν μιας συμφωνίας ε, που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των κοινωνικών στρωμάτων όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Ε, οι, μόνο οι μεγάλες εταιρείε βγάζουν κέρδη από αυτό. Ε, πίσω από τα διαμάντια που εισάγουμε από το Μποτσουάν, από το πετρέλαιο της Αγγόλας ε, ή από τα μέταλλα και τους πολύμους λίθους της Ναμίμπια βρίσκονται τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε 31 εκατομμύρια και εξήγαγε 33 εκατομμύρια θετικός κατά 2 εκατομμύρια ο ισολογισμό. Όλα αυτά πήγαν στις τσέπες ε, των επιχειρήσεων ε, που ε, εισάγουν αυτά, αγοράζουν αυτές τις πρώτες σύλλε σε χαμηλή τιμή. Κυρία Τζουφρίντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα αυτή τη συμφωνία. Καταψήφισα τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιε ε, χώρε τη ε, Αφρική, μεταξύ αυτών και η Νότια Αφρική, γιατί αυτό θα ήταν άλλο ένα πλήγμα για την ε, γεωργία, κυρίω τη νότια Ευρώπη. Τα προκυπευτικά μα τα πορτοκάλια της περιοχής μου που είναι τα καλύτερα. με λοιπόν αντίθετη γιατί θέλω να πω φτάνει. Φτάνει πια σε εμπορικές συμφωνίες που οδηγούν στην εκμετάλλευση, στο να είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε εδώ προϊόντα χωρίς καν να μπορούμε να τα ελέγξουμε, χωρίς να γίνουν φυτογειονομικοί έλεγχοι. Λέω λοιπόν φτάνει στην ε, Γεωργία ε, και λέω επίσης φτάνει στο μονοπόλιο γιατί η Επιτροπή τελικά καταλήγει στο να συνάπτει συμφωνίες ε, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη της τι επιπτώσεις έχουν όλες αυτές οι συμφωνίες στις τοπικές αγορές. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει κάτι, τότε οι δική μας οι γεωργοί είναι να φέρουν το βάρος λανθασμένων αποφάσεων. Begin, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ εμείς δηλαδή από τη, τα, τους πέντε αστέρες ε, καταψηφίσαμε γιατί η συμφωνία αυτή υποτίθεται είναι μια συμφωνία για να βοηθηθεί η Αφρική αλλά είναι μια ε, συμφωνία η οποία θα ανοίξει κατά 86% της ε, αγορές της Αφρικής. Αυτό είναι απαράδεκτο. Χάνονται πάρα πολλά κονδύλια. Και παράλληλα για μας η πρώτη συνέπεια είναι ότι θα έχουμε πορτοκάλια από την Νότια Αφρική Υπότιτλοι AUTHORWAVE όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται η συμφωνία. Εμείς θέλουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνία των πολιτών δεν περιλαμβάνεται. Αυτή λοιπόν η συμφωνία μπορεί πολύ άνετα να οδηγήσει στη διάλυση ε, γιατί θεωρείται και η Νότια Αφρική ότι είναι μια μικρή χώρα. Επίσης αναγκάζουμε τους εταίρους μας να υπογράψουν κάτι χωρίς οι δικοί τους οι βουλευτές να έχουν το χρόνο να διαβάσουν το κείμενο που υπογράφουν. Και αν δεν υπογράψουν ε, θα τους τιμωρήσουμε με δασμούς ε, αλλά ε, φαίνεται ότι με την Αφρική πάντα αυτό κάναμε και υποτίθεται έχουμε και δημοκρατία. Ωραία, θα περάσουμε στις προτάσεις ε, στα σχέδια ψηφίσματος. Πρώτο θέμα η Πολωνία. Ο κύριος Χάναν δεν είναι στην αίθουσα. Γεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την ε, αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δούμε λιγάκι ε, το νόημα του ψηφίσματος θα διαπιστώσουμε ότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Μεταξύ φίλων είναι καλό να λέει κανείς την άποψή του αλλά και να επισημαίνει και λάθη. Και μεταξύ φίλων είναι επίσης σημαντικό να τηρούνται οι συμφωνίες. Ε, και γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, με το ψήφισμα αυτό, αυτό ζητάμε, ε, πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί το ψήφισμα και με τον τρόπο αυτό μπορεί να έχουμε και ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, συνάδελφοι. πρόκειται για μία ε, παρέμβαση ε, στις εσωτερικές υποθέσεις. Παιδιά, ε, της εθνικής κυριαρχίας ε, των κρατών μελών υπάρχουν αυξανόμενες υποψίες από πλευράς ε, των πολιτών ε, κατά των ηθινόντων. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις ε, που θα υποστηρίξουν την επικουρικότητα, την εθνική κυριαρχία και την αυτοδιάθεση. Είμαστε μάρτυρες ενός, μιας εξέλιξης που συζητήθηκε στο Συμβούλιο. Είναι κυρίαρχο ε, κράτος ε, η Πολωνία. Διακόπτει ο πρώτος. Ναι, ευχαριστώ. Ε, καταψήφισα το ψήφισμα παρότι είμαι πολέμιος ε, το, της τωρινής κυβέρνησης, όμως οποιοδήποτε έξωθεν πίεση υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και νομίζω ότι με αυτό το ψήφισμα θα υποστηρίξουμε τελικά την κυβέρνηση, θα γίνει πιο δημοφιλής ακόμη. η τωρινή πολωνική κυβέρνηση κατακρίνεται μέσα σε αυτό το ψήφισμα και προηγούμενη κακή ήταν και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα στις εκλογές. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη δημοκρατία στην Πολωνία και προσπάθει να δει πώς λειτουργεί. Ε, είναι γκροτέσκο. Κοιτάξτε την Αυστρία. Εδώ και μήνες δεν διεξάγονται προεδρικές εκλογές ε, ε, ενώ θα έπρεπε. Δεν τα καταφέρνουν. Ε, ο ορισμός οικογένειας, οι μειονότητες, όλα αμφισβητούνται. Βλέπετε ότι στην Γαλλία πολλά μεγάλα κόμματα δεν έχουν προσώπηση στο κοινοβούλιο. Ε, και μιλάμε μόνο για την Πολωνία. Για το πώς εκλέγουμε τον πρόεδρο. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση για την Ισία. Ο κύριος ε, Ανάν δεν είναι εδώ. Περνάμε το, στην κυρία Φορέντσα. Μικρόφωνο παρακαλούμε θα ήθελα να εξηγήσω γιατί δήλωσα αποχή για αυτή την εκθεσία, όχι διότι δεν εκτιμώ τις ε, προσπάθειες που καταβάλει ο εισηγητής κ. Καστάρντο, αλλά διότι πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία, ε, κυρίως ε, σε σχέση με αυτό που θεωρείται η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των Τινησίων. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε εγκαταλείψει τους Τινήσιους ε, υπάρχει μια πολιτική ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών ε, που δεν βοηθάει όμως τους τινήσιους, δεν βοηθάει ε, τους μικρούς γεωργούς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί όσον αφορά το θέμα της αύξησης των ποσοστώσεων ελαιολάδου όπως προβλέπεται στις ελεύθερες εμπορικές ανταλλαγές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τινησία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει κυρίως να στηρίξουμε την Τινησία στο θέμα του χρέους που πλήττει ε, την κυβέρνηση και τους πολίτες. Κύριε Μακοβέη, πέντε χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη ε, η κατάσταση στην ε, την Ισία είναι μάλλον υποδειγματική. Ένα παράδειγμα πρέπει να ακολουθεί και από άλλε χώρε. Η Τινησία αυτή τη στιγμή αποτελεί ε, σπίτι ενός καταφύγιου, δηλαδή ενό εκατομμυρίου Λίβιων που έχουν ξεφύγει από τον πόλεμο. Χρειάζεται λοιπόν ένα πραγματικό πρόγραμμα Marshall για να παγιωθεί η δημοκρατία εκεί. Μόνο με μια ισχυρή δημοκρατία, ένα ισχυρό κράτο στην Τινησία μπορούμε να έχουμε ελπίδε για μια σταθερή περιοχή, περιφέρεια ε, στο σύνολό της. Χρειάζεται μια ανεξάρτητη αρχή για τις κρατικές προμήθειες και για την παρακολούθηση της λειτουργίας ε, του κράτους. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει αποτελεσματικότητα και διαφάνεια και βέβαια οι επενδυτές θα υποφεληθούν και θα δώσουν το παρόν. Η πρόταση ε, προτείνει τη δημιουργία ενός σημείου επαφής μέσω Eurojust με την Τινησία πολύ θετικά όλα αυτά. Ελπίζω ότι τα πράξεις θα ακολουθήσουν τα λόγια. Ευχαριστώ κ. Μάουλου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση ε, λόγω της φύσης της συμφωνίας ε, γιατί είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα η οποία πράγματι ξεκίνησε τις μεταρρυθμίσεις Μπορεί λοιπόν αυτό το μοντέλο της Τινησίας να εφαρμοστεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό. Να εξασφαλίσουμε ότι οι περισσότεροι νέοι στην Τινησία θα έχουν ε, ένα μέλλον, ε, να μην ε, ενδώσουν στον προσελητισμό που ασκείται και σε αυτό το κράτο, αλλά κυρίως την, την Ισία μπορούμε να τη θεωρούμε ένα εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ολοκληρωθεί η δημοκρατική διαδικασία ε, με τις σχέσεις με την Ιταλία, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισία είναι πολύ καλές και μπορέσαμε εμεί λοιπόν να ε, σταθεροποιήσουμε, να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η χώρα θα έχει τις βέλτιες δυνατές συνθήκε που μπορούν να επιτύχει. Κιουτσούκ, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ υποστήριξα την έκθεση διότι δεν, ε, η Τινησία δεν είναι χώρα μόνο όπου άρχισε η Αραβική Άνοιξη, αλλά επιδόθηκε ε, και κατοχυρώθηκε το κράτος ε, του δικαίου και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, ε, λειτουργεί εύρυθμα η κοινωνία των πολιτών. Παρόλα αυτά υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Ε, αστάθεια σε κάποιες περιοχές, μεγάλη απειλή από τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό πλήττει φυσικά την τουριστική βιομηχανία. Χρειάζεται την βοήθειά μας προς τον εκδημοκρατισμό, την καλή διακυβέρνηση η την Ισία και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, κάτι που είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ισία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε βοήθεια για τα προγράμματα από Είναι καλύτερη η πρόληψη για την τρομοκρατία. Ευχαριστούμε. Ο ε, πως Πισίλα αποσιάζει. Έκθεση μπάλας. Είναι η σειρά του κυρίου Ανάν και πάλι, αλλά δεν είναι. Εδώ απουσιάζει Φορένζα. Θα ήθελα να, ευχαρισ... να εξηγήσω για ποιο λόγο υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Είναι ένα πρώτο βήμα στον αγώνα κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Φυσικά είναι ένα πρώτο βήμα και υπολείπεται μακρύς δρόμος για να κερδίσουμε σε αυτόν τον αγώνα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Είναι ε, ε, μια κατάσταση άγριας, ξέφρενης ε, παγκοσμιοποίησης που οδηγεί σε μια έκρηθμη απελευθέρωση πλήττοντας ε, τα εργασιακά δικαιώματα. Πρόκειται για έναν αγώνα προς τα κάτω. Αυτή είναι η ρίζα του κοινωνικού ντάμπινγκ και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε θεσπίσει τα πρότυπά μας ε, για το εργατικό δίκαιο συμπληρώνοντας την εθνική νομοθεσία ε, χωρίς να ξεχνάμε και το θέμα της ηθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγος Φαρμέχου η χειροτέρευση των ρεσιακών σχέσεων και των κοινωνικών δικαιωμάτων εξαιτία του κοινωνικού ντάμπινγκ είναι το θεμελιώδε ε, πρόβλημα τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συνεχή διάβρωση εδώ και δεκαετίε που ε, φτωχοποιεί του εργαζόμενου στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει τα εργαλεία για να καταπολεμήσει αυτή την πρακτική, αλλά οι οδηγίε που εγκρίνονται, όπω για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών, δεν εφαρμόζονται ή ε, όπως έγινε με την ε, νομοθεσία των ε, μετακινούμενων εργαζόμενων ε, διαλύονται το περιεχόμενο τους χειροτερεύει με το χρόνο. Θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα και οι ποινές που έχουν προβλεφθεί. Να καταπολεμηθούν οι εικονικές έδρες, οι εικονικές επιχειρήσεις και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Το απαιτούν οι νόμοι και οι βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υποτιμάται κάθε μέρα που περνάει. Ε, μόνο έτσι θα ε, περασπίσουμε τη μια δημοκρατική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ παράθυρα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και η αποδυνάμιση των ε, συλλογικών συμβάσεων έχουν τύχει εκμετάλλευση από τους εργοδότες και δημιουργείται ε, αθέμητος ανταγωνισμός. Ε, η ξενοφοβία, το μίσος για τους μετανάστες επιδεινώνονται για αυτό το λόγο. Πολλοί από τους δικούς μου ψηφοφόρους φοβούνται ότι απειλείται η ζωή τους και η ευημερία τους με την ε, εισαγωγή εργατικού δυναμικού και με άλλους τρόπους ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπ και γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ σημαντική αυτή η οδηγία, την υποστήριξα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία στο ίδιο γεωγραφικό σημείο και σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα σήμερα, οι συνέπειε για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καταστροφικέ μακροπρόθεσμα και θα μπορούσαν να υποσκάψουν ακόμα και την ίδια την ύπαρξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Κόρβιν Μικέ. Καταψήφισα προφανώς αυτή την έκθεση αυτό το ψήφισμα διότι θα δημιουργήσει ένα καινούριο εργαλείο ε, χωρίς λόγο. είναι ένα εργαλείο το οποίο θα περιορίσει την ε, ελεύθερη πρόσληψη. Ε, θα απαγορεύσει τους εργαζόμενους να μπορούν να πουλήσουν το κοινωνικό τους πλεονέκτημα και να λάβουν χρήματα ως αντιστάθμισμα. Ε, είναι προφανές ότι κάποιοι συνάδελφοι ξέρουν καλύτερα τι χρησιμεύει και τι είναι αυτό που θέλουν οι εργαζόμενοι. Η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο ζητάει περισσότερους ελέγχους και λιγότερη ελευθερία. Ακόμα και επί Στάλιν υπήρχαν διαφορετικές ρυθμίσεις σε διαφορετικές χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Γιούρεκ. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι είναι Ευρώπη των Εθνών θα έπρεπε να στηρίξουμε μια ενιαία αγορά και όχι να την περιορίζουμε. Θα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις χώρες μας. Ε, επί κομμουνισμού κάποιες χώρες ε, αποσπάστηκαν από την Ευρώπη, δεν θα πρέπει να το επιστρέψουμε και δεν θα πρέπει να μειώσουμε την ελευθερία που έχουν, να περιορίσουμε την ελευθερία που έχουν οι πολίτες τους να εργάζονται. Εμείς στην ε, Πολωνία γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μας βεβαίωσαν ότι θα μπορούσαμε να λειτουργούμε σε μια νέα αγορά γνωρίζουμε τον ανταγωνισμό και θέλουμε να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό μας, όχι να τον περικόψουμε. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν. Στήριξα αυτή την έκθεση για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Και μια ακόμα φορά σήμερα ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, ανακοίνωσε ίδια αμοιβή για την ίδια δουλειά στον ίδιο γεωγραφικό τόπο και χαίρομαι γι' αυτό. Ίδια αμοιβή για ίδια εργασία στο ίδιο σημείο είναι σημαντικό για αυτή την Κομισιόν και νομίζω ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες συμμερίζονται αυτή την άποψη. Είναι κέριο θέμα, ε, θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση στήριξα το, την πρόθεση των ελάχιστων ε, εθνικών μισθών ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε ελάχιστο μισθό και θα πρέπει αυτός ο καθορισμός να γίνεται σύμφωνα με τις ε, εθνικέ παραδόσει και τι εθνικέ ρυθμίσει. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι αξιοπρεπεί μισθοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή και η κοινωνική συνοχή είναι το αντίδοτο του κοινωνικού ντάμπινγκ. Το κοινωνικό ντάμπινγκ υποσκάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε μέχρι τις 3.